Ζητώ συγγνώμη, συνάδελφοι, συνάδελφε, που άργησα. Λοιπόν, ξεκινάμε το σημείο 13 παρουσίαση από την Κομισιόν μιας πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου <clears throat> για το κεκτημένο Σέγγεν ε, στην Δημοκρατία της ε, Κροατίας. Ο κύριος Νέλο έχει τον λόγο και ζητώ και πάλι συγγνώμη που άργησα. Α, συγγνώμη, όχι, πρέπει να ακούσουμε την Κομισιόν πρώτα. Ποιον, θα ακούσουμε τον κύριο Κλήρωτ. Ωραία, Κομισιόν. Thank you, uh, Mr. Chair, um, and good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Ευχαριστώ. Βίλα Κλάρχοντ, δουλεύω στη Γενική Διεύθυνση HOME, ε, στην, ε, στο τμημα ΜΗΤΡΙΑ που ασχολείται με τα συστήματα πληροφορική ε, του Σέγγεν. κυρίω. Να σας εξηγήσω λιγάκι το πλαίσιο της πρότασης και να πω και δύο λόγια για το πλαίσιο και τις επιπτώσεις. Καταρχά να σας εξηγήσω ότι αυτή η πρόταση συνδέεται με την συνεχιζόμενη διαδικασία αξιολόγηση Σέγγεν τη Κροατία, Ο στόχος της αξιολόγηση Σέγγεν γενικά, αλλά και ειδικά για τη Κροατία, είναι να ε, επαληθεύσουμε με βάση το 4-2 της πράξης προσχώρησης της Κροατίας, εάν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ε, πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν. Και μετά από την ε, επιτυχή αξιολόγηση της Κροατίας, το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να λάβει μια απόφαση για την πλήρη εφαρμογή όλων των τμήματων του κεκτημένου του Σέγγεν στην Κροατία. Η αξιολόγηση της Κροατίας ξεκίνησε το 2016 μετά τη δήλωση της Κροατίας ότι είναι έτοιμη να αξιολογηθεί από την Κομισιόν το 2015. Και η αξιολόγηση καλύπτει διάφορες πτυχές. Τον κώδικα θεωρήσεων, την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, την ε, αστυνομική συνεργασία, την προστασία των δεδομένων και τη λειτουργία του ΣΥΣ, του Συστήματος ε, Πληροφόρησης Σέγγεν. Αυτή η τελευταία αξιολόγηση του ΣΥΣ δεν έχει λάβει ακόμα χώρα, δεν έχει γίνει επίσκεψη ακόμα, γιατί μπορεί να γίνει μόνο αυτή τη στιγμή στο σύστημα γίνει λειτουργικό στην Κροατία γιατί το σύστημα πληροφοριών του ΣΕΝΚ είναι ένα σύστημα πληροφορική, ε, γίνεται επιχειρησιακό. Επομένω, οι επιχειρησιακέ και τεχνικέ λειτουργίε μπορούν να αξιολογηθούν, οι λειτουργικέ του, α πούμε, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, μόνο αυτή τη στιγμή αρχίσει να τρέχει. Το θέμα της πρότασης λοιπόν είναι να επιτρέψουμε την βαθμιαία ε, εφαρμογή του συστήματος ΣΥΣ στην Κροατία και όπως εξηγεί και η επεξηγηματική έκθεση το μνημόνιο αυτό, η Κροατία πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ε, ούτως ώστε το Συμβούλιο να μπορέσει να λάβει αυτή την απόφαση, η προστασία των δεδομένων. Και η αξιολόγηση αυτή ε, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2016. Η Κροατία επίσης, τεχνικός πώς είναι έτοιμη να συνδεθεί με το ΣΥΣ, έχει το δικό της εθνικό σύστημα, έχουν ένα γραφείο ΣΥΡΕΝΕ και έχουν ε, τσεκάρει την δυνατότητα επικοινωνίας με τα άλλα γραφεία ΣΥΡΕΝΕ και είναι οκ. Προτείνεται λοιπόν το Συμβούλιο να αποφασίσει σε δύο ημερομηνίε που αναφέρονται στην πρόταση, στο άρθρο 1 παράγραφος 2 την ημερομηνία από την οποία ε, τα δεδομένα του ΣΥΣ που έχουν ε, δημιουργηθεί από τα άλλα κράτη-μέλη μπορούν να δοθούν στην Κροατία. Και η δεύτερη ημερομηνία είναι η ημερομηνία από την οποία και, μετά μπορεί η Κροατία να αρχίσει να δημιουργεί τις δικές της, τα δικά της alert. Και, θα, και υπάρχει στην παράγραφο 1 και 3 του άρθρου 1 το στοιχείο αυτό. Μια και το Συμβούλιο επίσης δεν έχει λάβει την τελική απόφαση για την πλήρη εφαρμογή όλων των στοιχείων του κεκτημένου ΣΕΝΚΕΤ που μπορεί να γίνει μόνο από την, ε, μετά την πλήρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της Κροατίας, θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για τη χρήση των δεδομένων ΣΥΣ από την Κροατία. Και αυτό αφού έχει να κάνει με την άρνηση εισόδου δηλαδή alert για αυτά τα θέματα, μέχρι εκείνη την ημερομηνία δηλαδή η Κροατία δεν θα μπορεί να βάζει ε, στο ΣΥΣ τέτοιου τύπου συστήματα, και θα, ε, δεδομένα μάλλον, και δεν θα μπορεί να αρνηθεί ε, την είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε alert τρι, ε, άλλων κρατών μελών. Αυτά εξηγούνται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1. Ευχαριστώ πολύ πριν πάω κύριε κύριο Μέλλο να ακούσουμε για τη Μαλτέζικη Προεδρία. Ο κύριος Κασέρη. So, honorable Αξιότιμα μελή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως εκπρόσωπος, ε, όπως είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, τα κράτη-μέλη με την Κομισιόν αυτή τη στιγμή αξιολογούν την εφαρμογή την εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν και την ορθότητά της σε διάφορους τομείς. Ένας από αυτούς είναι η προστασία των δεδομένων και αποτελεί προϋπόθεση ώστε η Κροατία να μπορέσει να ξεκινήσει την ανταλλαγή επιπρόσθετων πληροφοριών και τη χρήση του ε, συστήματος πληροφοριών Σέγγεν. θα, πω, θα εξετάσω τα ίδια με τα οποία, στα οποία αναφέρθηκε η Κομισιόν με κίνδυνο να επαναλάβω. Η Κομισιόν ε, υιοθέτησε την έκθεση αξιολόγηση, έχει επαρκή προστασία δεδομένων η Κροατία, διαπίστωσε και τώρα το Συμβούλιο θα κάνει τα επόμενα βήματα, θα προχωρήσει στα σχέδια αποφάσεων ε, που ήδη εξετάζει Όλα αυτά θα γίνουν βάσει του άρθρου 4.2 της ε, πράξης προσχώρηση της ε, Κροατίας ε, και 1η Ιανουαρίου ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου μέχρι την Ολομελία του Μαρτίου, αν είναι αυτό δυνατόν. Ο λόγος για αυτή την πίεση ήταν να μην αλλάξει το χρονοδιαγράμμα των σημερινών αξιολογήσεων Σέγγεν. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην αξιολόγηση αυτή που προβλέπεται να λάβει χώρο στον Ιούλιο του 2017 θα θέσει κίνδυνο την πλήρη προσχώρηση στο Σέγγεν. Την άρση δηλαδή των ελέγχων εσωτερικών συνόρων, η οποία πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Ειδικότερα διότι η Κροατία τεχνικώς είναι έτοιμη να προσχωρήσει στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. έχει στο το γραφεία τις ε, απαραίτητες διαδικασίες ήδη από το καλοκαίρι του 2016. Η θέση σε λειτουργία του συστήματος ε, ε, στην Κροατία είναι σημαντική και στο πλαίσιο του ΣΥΡΕΝ, διότι θα διευκολύνει τη συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Κάποιε πτυχέ τη συνεργασία ε, υπάρχουν ήδη, όπω η χρήση Ευρωπα... τη ε, απόφαση πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, αλλά η Κροατία δεν μπορεί ακόμα να χρησιμοποιήσει το ΣΥΣ για alerts ε, βάσει ευρωπαϊκών ενταλμάτων για απελάσει. Προ το παρόν είναι αναγκασμένη να χρησιμοποιεί τη δικά τη συστήματα, όπως και για εκδόσει επειδή δεν έχει τη σύνδεση με το ΕΣΕ, σε δύο-τρει μήνε. Ε, για δύο-τρει μήνε η Κροατία θα χρειαστεί να φορτώνει τα δεδομένα και να ελέγξει τη λειτουργία του συστήματο ε, πριν από την αξιολόγηση του συστήματο πληροφοριών Σέγγεν. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο θα ήθελε να έχει τη δική σα γνωμοδότηση το συντομότερο δυνατόν κατά προτίμηση μέχρι τα τέλη του μήνα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σε ευχαριστώ. Μετά από τα όσα είπατε, το Κοινοβούλιο μπορεί να δεχτεί να απορρίψει το κείμενο και δεδομένης ε, της ε, γρηγορής ε, έγκρισης η προθεσμία είναι αύριο Παρασκευή 10 στις 4 το απόγευμα και μετά θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 7 Μαρτίου και μετά θα πάμε στην πρώτη ολομέλεια του Απριλίου. Λοιπόν, μετά από αυτά θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή να κάνει την παρουσίαση του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά αν δεν σας πειράζει. Το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν δημιουργήθηκε για να υπάρχει εσωτερική ασφάλεια και έλεγχος των εξωτερικών συνόρων στις ε, χώρες Σέγγεν και αφορά ανταλλαγή δεδομένων Σέγγεν για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ζώνης Σέγγεν. Τώρα, το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει μια απόφαση για το εάν αυτά ισχύουν στην ε, Κροατία μετά από τα... την λήψη των τεχνικών και νομικών μέτρων. Όταν μιλάμε για τις ε, τεχνικές ε, διατάξεις, η αξιολόγηση φαίνεται ότι είναι θετική και θεωρείται ότι η Κροατία πλήρει τα κριτήρια και παρέχει το απαραίτητο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα. Για την επιχειρησιακή πτυχή συλλογής ε, πληροφοριών μεγάλης κλίμακας. Ε, υπάρχουν και τα τεχνικά κριτήρια. Η αξιολόγηση της ε, Κροατίας για το σύστημα θα γίνει όταν ενταχθεί η χώρα στο σύστημα Σέγγεν και στηρίζουμε την απόφαση του Συμβουλίου και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών έτσι θα πούμε, να βελτιωθεί μπορεί η ασφάλεια στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και προφανώς ε, στην προτεραιότητα της ε, πολιτικής μου μας. Ε, αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. ή άλλη βουλευτής ή παρούσα θα ήθελε να πει κάτι και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους και το προσωπικό για την καθυστέρηση μου. Κυρία Σίπελ, ναι, ευχαριστώ. Δεν ε, ήθελα να παρέμβω, ήθελα απλά να ακούσω και να ενημερωθώ, αλλά θα ήθελα να κάνω μια πολιτική δήλωση γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι προφανώς παρά το ότι και άλλα κράτη-μέλη πληρούν τα τεχνικά κριτήρια δεν ε, είναι όλα τα κράτη-μέλη μέρος του συστήματος ε, πληροφοριών Σέγγεν. Οπότε δεν πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά στα κράτη-μέλη. Και αν η Κροατία πληρεί τα κριτήρια βεβαίως ε, να γίνει μέλος του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν, αλλά εγώ δεν μπορούσα παρά να μη διάσω όταν άκουσα ότι η Κομισιόν συμφωνεί ε, με το θέμα της προστασίας δεδομένων και μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί έχω και κάποιες εμπειρίες σχετικά με την προστασία δεδομένων ε, όταν λέει έχει πει η Κομισιόν τα ίδια πράγματα και για άλλες τρίτες χώρες αλλά τέλος πάντων σήμερα ήρθα κυρίως για να ακούσω και εάν τα κατήρια πληρούνται βεβαίως η χώρα να γίνει μέλος του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν. Σας ευχαριστώ που ε, έχουμε συζήτηση πλέον με την δική σας την παρέμβαση. Κύριε Μέλο, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, όχι. Ε, πληροφοριακά να σας πω. Η ψηφοφορία στις 22 Μαρτίου στην Επιτροπή και σύμφωνα με τον κανονισμό τροπολογίες θα γίνουν δεκτές μόνο εάν διαφωνούν με την ε, σύσταση του εισηγητή και δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το αυτόματο σύστημα κατάθεσης τροπολογιών γιατί δεν στηρίζει την διαδικασία αυτή της ε, διαβούλευσης. Οπότε πρέπει να στείλετε κλασικά ειδοποίηση στην γραμματεία, αν με ακούει ακόμα κανείς και κύριε Μέλο, σας ευχαριστώ και για την υπομονή σας. Και ευχαριστώ και την κυρία Σίπελ, η οποία επισήμως πλέον πρέπει να είναι το μέλος της Επιτροπής με την ε, καλύτερη προσέλευση. Τουλάχιστον όσο καιρό είμαι εγώ εδώ. Σας ευχαριστώ και τελειώσαμε. Άρα και με την συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δεν συνηθίζουμε να έχουμε μισά ώρες συνεδριάσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.